Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές μου ανακοίνωσαν ότι οι βουλευτές Αναστάζε, Κορλάτεν, Φίλιπ, Ιακομπρίτζη, Νέσιφορ, Οπρέα και Πόπα εκλέχθηκαν ως μέλη του Ρουμανικού Κοινοβουλίου. Ο, ο πρόεδρος είπε κατά λάθο του Ρωμαϊκού Κοινοβουλίου και τώρα το διορθώνει. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού για τις ε, άμεσες εκλογές για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού μας διαπιστώνω την απελευθέρωση των εδρών αυτών από 19 Δεκεμβρίου 2008. Οι Ρουμανικές αρχές μου ανακοινώνουν εξάλλου ότι από 22 Δεκεμβρίου 2008 έχουμε τους εξής ο κύριος Άντριαν Μανώλη αντικαθιστά την κυρία Αναστάζη, ο κύριος Μάτουλα την κυρία Γιακοπρίτσι, ο κύριος Κάλιν Τσιρίτα την κυρία Πόπα, ο κύριος Αλεξάνδρου Ναζάρε τον κύριο Φίλιπ και ο κύριος Ντάνιελ Πέτρου Φουνέριου τον κύριο Οπρέα. Αντικαθιστούν λοιπόν τα νέα αυτά μέλη, τα αποχωρήσαντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τους εύχομαι το καλώς ορίσατε μαζί με τα συγχαρητήριά μου. Οι αρμόδιες φιλανδικές αρχές μου ανακοινώνουν ότι η κυρία Εύαρητα Σίτονεν καταλαμβάνει την έδρα της κυρίας Κάουπη από 1η Ιανουαρίου 2009 και γίνεται μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού, τα νέα αυτά μέλη και εφόσον οι εντολές τους δεν έχουν εξεταστεί ή εφόσον δεν έχει ε, υπάρξει κρίση επί ιασδήποτε ενστάσεως αναλαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν γραπτή δήλωση σχετικά με το ότι δεν διατηρούν κανένα αξίωμα το οποίο να είναι ενδεχομένως ασυμβίβαστο με τα καθήκοντα του Ευρωβουλευτού. Μετά από ε, πρόταση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Ρόμπερτ Άτκινς δεν, δεν είναι πλέον μέλος της Επιτροπής μεταφορών. Η διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίασή της 8 Ιανουαρίου 2009 και σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού 45-2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και μετά από τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής